Ευχαριστώ. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις και για το γεγονός ότι μου δώσετε τη δυνατότητα να απαντήσω. Ευχαριστώ και τον κύριο Γιούγκερ που μου έδωσε τη δυνατότητα να βρίσκομαι εδώ. Επιτρέψτε μου να σας πω δύο λόγια παραπάνω για το όραμα της ε, Ενεργειακής Ένωσης και να σας δώσω και κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Έχουμε περιέλθει σε μια κατάσταση η οποία επιβάλλει ε, να αναλάβουμε δράση. Μετά το 2009 δεν έγιναν αρκετά για να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού. Πρέπει να έχουμε μία ανθεκτική ενεργειακή ένωση με το βλέμμα στο μέλλον. Και η στόχοι δηλαδή μία ε, κλιματική πολιτική με το βλέμμα στο μέλλον είναι σαφής. Κυρίως η στόχοι του 2020. 20% μείωση των ε, αερίων του φαινομένου θερμοκηπίου, 20% ε, ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 20% μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Οι στόχοι αυτοί θα έχουν συνέχεια τους στόχους για το 2030. 30% μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να υλοποιήσουμε προγράμματα μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης που θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε την περιβόητη πράσινη οικονομική ανάπτυξη. Και επίσης 27% ε, τουλάχιστον ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και ο στόχος ο οποίος ανέφερα και προηγουμένως για το 2050 και θεωρώ ότι θα έχουμε και υποστήριξη από τις πόλπες χώρες εταίρους, επ' αυτού είναι η μείωση κατά 80% των εκπομπών. Τα βασικά στοιχεία της Ενεργειακής Ένωσης στοιχεία τα οποία προέκυψαν και από την σημερινή συζήτηση είναι καταρχάς καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε καλύτερες υποδομές, καλύτερη διασύνδεση, μια ε, πιο ισχυρή οικονομική αγορά που θα μας επιτρέψει να δώσουμε κίνητρα για ανταγωνιστικότητα που είναι πολύ σημαντική και για την ε, βιομηχανία αλλά και για τους πολίτες. Στο παρελθόν είχαμε μια οικονομία υψηλής κατανάλωσης άνθρακα. Το πέρασμα στην οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα θα μπορέσουμε να το κάνουμε ε, μέσω ε, ενεργειακής αποδοτικότητας και μέσω αυτών των στόχων θα καταφέρουμε να μειώσουμε και την εξάρτηση από τις εισαγωγές. Και φυσικά το κερασάκι στην τούρτα θα πρέπει να ενισχύσουμε την κοινή μας δράση ενώπιον των διεθνών μας εταίρων. Όσο μεγαλύτερη βαρύτητα Όσο μεγαλύτερη ισχύ ε, έχουμε τόσο καλύτερο και αυτό φυσικά θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε εάν μπορούμε να δράσουμε από κοινού και αν μπορούμε να διασφαλίσουμε και μία κοινή θέση. Αυτό το οποίο αποτελεί για μένα προτεραιότητα, εάν μου δώσετε το χρήσμα, θα ε, είναι να καθορίσω με τους συνεργάτες μου ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης. ένα σχέδιο για το μέλλον για το ενδεχόμενο έλλειψης φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Οι συνεργάτες μου ήδη ετοιμάζουν το σχετικό έγγραφο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο ε, προσεχώς και είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι υπάρχει όραμα, υπάρχουν οι στόχοι και έχουμε ξεκινήσει μία άγουσα η οποία θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε το στόχο μας. Ευχαριστώ κυρία Αλένκα Μπράτουσεκ, υποψήφια αντιπρόεδρε και επίτροπε. Ευχαριστούμε για την καταληκτική αυτή η δήλωση. Ευχαριστώ τους συναδέλφους από τις δύο επιτροπές, όπως επίσης και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κοινής Γνώμης, είτε όσους παρίστανται, αλλά και αυτούς που μας παρακολουθούν μέσω διαδικτύου. Θα ήθελα να σας δώσω τελικές πληροφορίες για την Επιτροπή Ήτρε. Σήμερα το βράδυ στις 8 θα γίνει συνεδρίαση συντονιστών, ενώ αύριο όλοι μας όλα τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε. Έχουμε την ακρόαση του κυρίου Γιούρκη Κατάινεν στις 10 το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάποιες επιπλέον πληροφορίες για τους συναδέλφους της Επιτροπής ΕΝΒΗ. Η συνεδρίασή μας για την εξολόγηση θα γίνει από τις 7.30 έως τις 9 σήμερα το βράδυ με τους συντονιστές και κατόπιν θα ξεκινήσει η κοινή συνεδρίαση ε, συντονιστών επιτροπών Ήτρε και Ένβη από τις 9 ως τις 10. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.